Wznawiam posiedzenie. Ogłaszam Άρχεται η συνεδρίαση. Συνεχίζεται η συνεδρίαση μετά την διακοπή 25 Νοεμβρίου του 2010. Έχετε το σχέδιο των πρακτικών. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Όχι, εγκρίνονται. Θα ήθελα να κάνω κάποιες προκατακτικές ανακοινώσεις πριν περάσουμε στις εργασίες μας. Η διάσκεψη των Προέδρων την περασμένη Πέμπτη έλαβε κάποιες αποφάσεις. Αύριο στις 4 η ώρα θα κάνουμε μία συζήτηση για την έκθεση της κυρίας Ιδονίας Ζενιέσκα και της κυρίας Τρίπελ για το νέο σχέδιο προϋπολογισμού του 2011. Έχει προγραμματιστεί η ψηφοφορία για την Τετάρτη. Δεύτερη ανακοίνωση, αύριο θα γίνει συζήτηση για τα αποτελέσματα της COP16, της διάσκεψης της Κανκούν για τις κλιματικές αλλαγές. Σημειώθηκε πρόοδος στην Κανκούν και ένα κλιμάκιο του Κοινοβουλίου φυσικά συμμετείχε στη διάσκεψη. Οι συνάδελφοι είναι σήμερα μαζί μας και από κοινού με την Επίτροπο θα συζητήσουμε τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε τελικά να αποβεί επωφελής η συμφωνία ε, και θα προετοιμάσουμε τη διάσκεψη στη Νότιο Αφρική. Ε, στις 21 Οκτωβρίου μάθαμε για το βραβείο Ζαχαρόφ, Ζαχαρόφ για την ελευθερία της σκέψης. Ο Γκυγέρμο Φαρίνιας κέρδισε το βραβείο Ζαχαρόφ. Δυστυχώς ο κύριος Φαρίνιας κολλείεται ε, για να μεταβεί στο Κοινοβούλιο και να παραλάβει αυτοπροσώπως ε, το βραβείο. Επέμεινα εγώ ίδιος ε, και έστειλα επιστολή στον κύριο Ραούλ Κάστρο. Προς το παρόν είναι αδύνατο να γίνει κάτι και λόγω του ότι ο κύριος Φαρένιας δεν μπορεί να μεταβεί στο Κοινοβούλιο, υποθέτω ότι η κυρία Άστον θα λάβει υπόψη την κατάσταση των και των σχέσεων που έχουμε με την Κούβα. Ευελπιστούμε ε, ότι θα μπορέσει τελικά να έρθει εάν φύγει τις προσεχείς ώρες ε, από την Κούβα θα μπορούσε να φτάσει εγκαίρος για την ε, απονομή. Κατόπιν ε, στις 13 ε, Δεκεμβρίου 81, πριν 20 χρόνια, κηρύχθη η πολιορκία στην Πολωνία και προσπάθησε η κομμουνιστική κυβέρνηση ε, να επιδείξει αλληλεγγύη Είχαμε πάνω από 100 θανάτους, πολλούς τραυματίες. Πέρασαν όλες αυτές οι δεκαετίες ε, και αποτείουμε φόρο τιμής για όσους αγωνίστηκαν για να ελευθερώσουν την Ευρώπη. Πέμπτη ανακοίνωση. Ε, δοθεί στη συμπεριφορά του κυρίου Μπλουμ στην ε, τελευταία σύνοδο Ολομέλειας και λόγω του ότι βάσει του άρθρου 9 και 153 του κανονισμού ε, δεν απολογήθηκε, ε, άρα αποφασίζω ότι για 7 ημέρες δεν θα λάβει την ημερήσια αποζημίωση στο Περντίεμ. Έχω ενημερώσει ε, προσωπικά και τον κύριο Μπλουμ για αυτή μου την απόφαση. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να σας ενημερώσω για την υπογραφή πράξεων βάσει της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Την Τετάρτη ο Πρόεδρος Συμβουλίου και εγώ θα υπογράψουμε μια δεκάδα τέτοιες νομικές πράξεις βάσει της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 74 του ιστορικού κανονισμού.